Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, υποψήφιο επίτροπο για την κλιματική δράση και την ενέργεια, κυρίον Μιγέλ Άρια Κανέτα, σε αυτή τη δημόσια ακρόαση που διοργανώνεται από κοινό από την Επιτροπή για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Επιστηστική Ασφάλεια και την Επιτροπή Βιομηχανίας ε, έρευνας και ενέργειας. If you wait, I'm going to explain. Μισό λεπτό, θα σας εξηγήσω. Μισό λεπτό. Ο Μιγγέλ Άριας Κανιέτε είναι αυτή τη στιγμή μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν ε, βουλευτής από το 1986 με το 1999 και ήταν πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, Αλίας από το 1995 στο 1997 και πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης από το 1997 έως το 1999. Στην Ισπανία ήταν επανειλημμένα γερουσιαστής και βουλευτής, υπουργός γεωργίας από το 2000 στο 2004 και Υπουργό Γεωργίας ε, Επιστημισμού και Περιβάλλοντος από το 2011-2014. Στην τελευταία του ιδιότητα εκπροσώπησε την Ισπανία στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη συναντήση κορυφή των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή στην Τόχα και την Βαρσοβία. Το χαρτοφυλάκιό του καλύπτει ε, ε, πολλά θέματα που είναι κεντρικά για την ε, λειτουργία των δύο επιτροπών μας. Όσον αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την οποία έχω την τιμή να, τις οποίες έχω την τιμή να προεδρεύω, εδώ και πολύ καιρό έχουμε δεσμευτεί για μια αποτελεσματική και φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα για να μειώσουμε ε, τις εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου και για να έχουμε μια βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη. Ανάμεσα στι νέε προτεραιότητες τι κύριε προτεραιότητά μα είναι να υπάρχει ουσιαστική ηγεσία τη Ένωση στι διεθνεί κλιματικέ διαπραγματεύσει εν ώψη τη συνάντηση κορυφή στο Παρίσι του 2015. Η σημασία να υπάρχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την ενέργεια, για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και η αναγκαιότητα να μεταρρυθμιστεί η αγορά ε, άνθρακα στην Ένωση και ιδιαίτερα το σύστημα ανταλλαγή ε, εκπομπών. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τι ε, κατευθύνε γραμμέ για την έγκριση τη Επιτροπή, το Κοινοβούλιο εκτιμά την ικανότητα των υποψηφίων επιτρόπων με βάση τις γενικές τους ικανότητες, τη δέσμευσή τους για τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και την προσωπική ανεξαρτησία. Επίσης, αποτιμά την γνώση τους του χαρτοφυλακίου και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Πριν την ε, ακρόαση, οι γραπτές απαντήσεις που μας έστειλε ο Επίτροπος έχουν διανεμηθεί. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου όλες οι άλλες ε, μεταφράσεις διανεμήθηκαν ε, στα μέλη σήμερα το πρωί. Πριν να σας παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η ακρόαση, θα δώσω το λόγο στον Σνάλφο Μπούζεκ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για την έρευνα, την, ένεργη, την βιομηχανία, την έρευνα και την τεχνολογία για τις αγωγικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, συνάδελφε Λαβία. Συμπροεδρεύουμε αυτή τη συνεδρίαση και θέλω να καλωσορίσω τον υποψήφιο επίτροπο Μιγέλ Άρια Κανιέτε που είναι ευρωβουλευτής άρα είστε σας στο σπίτι σας και καλωσορίζω και όλους τους συναδέλφους από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και την Επιτροπή Βιομηχανίας. Συνεργαζόμεθα πολύ. Πρέπει να συνεργαστούμε και συνεργαζόμεθα. Ε, όταν ε, πρώτο είναι Ευρωβουλευτής ήμουν ε, μέλος και των δύο επιτροπών αυτών για πέντε χρόνια και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας, μη κυβερνητικών οργανώσεων εταιριών, κρατών μελών, και επειδή είναι δημόσια ακρόασή μας και μεταδίδεται στο διαδίκτυο από τον ιστότοπο του Κοινοβουλίου ζωντανά. Λοιπόν, η Επιτροπή μας είναι αρμόδια για την ενεργειακή πολιτική, που είναι πολύ σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου του μέλλοντος επιτρόπου. Έχουμε τρία ενδιαφέροντα θέματα. Ενέργεια, ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας και νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα τρία θέματα είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με τα θέματα του κλίματος. Είναι αρμοδιότητα της Ήτρα. καθώς και άλλα. Η εσωτερική αγορά ενέργειας, η ασφάλεια της ε, προμήθειας ενέργειας, η προώθηση της ε, διασύνδεσης ε, των δικτύων, προώθηση των διευρωπαϊκών δικτύων, έρευνα ιδίως στον τομέα της ενέργειας, ενεργειακή ένωση. Όλα αυτά είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ήτρε. Άρα μας ενδιαφέρει πολύ να ακούσουμε τον κύριο υποψήφιο επίτροπο για το πώς προτίθεται να επιτελέσει το έργο αυτό. Και τέλος, η ενεργειακή μας πολιτική βασίζεται στο λεγόμενο τρίγωνο ενέργειας. Ασφάλεια, λογικές τιμές, προσιτές τιμές και περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω δράσης για το κλίμα. Χρειαζόμαστε μια σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των στόχων. Αυτή η ισορροπία θα είναι βασικό καθήκον του Επιτρόπου για την κλιματική δράση και την ενέργεια. Και υπάρχει μια νέα ευκαιρία για μια νέα αρμονία μεταξύ των μέσων και στόχων μας. Και τέλος, είναι ουσιώδες για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας με βιώσιμο τρόπο, αλλά επίσης για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ενεργειακές κρίσεις και για να σταματήσει η ενέργεια να αξιοποιείται ως μέσο πολιτικής πίεσης, ως όπλο. Πολλούς στόχους λοιπόν έχουμε ενώπιόν μας για την επόμενη πενταετία και θα συνεργαστούν οπωσδήποτε και οι δύο επιτροπές και αυτή η πρώτη ε, κοινή συνεδρίαση είναι μία απόδειξη της ε, θέλησής μας να συνεργαστούμε. Παρακαλώ κύριε Λαβία, σας δίνω και πάλι το λόγο. Έχει ζητηθεί διαδικαστικό. Με συγχωρείτε, αλλά πριν προχωρήσουμε στην ακρόαση, έχω ένα διαδικαστικό από πλευρά της Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Τι τελευταίε ε, τρεις ώρες ο επίτροπο κ. Κανιέτα άλλαξε τρει φορέ τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δημιουργεί σύγχυση για το εάν η νομική επιτροπή αποτίμησε σωστά εάν συμμορφούνται προ τι υποχρεώσει του. Γι' αυτό ζητώ επισήμω από εσά του δύο προέδρου των δύο επιτροπών ο κύριος Λαβία, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι διαδικαστικό. Είναι διαδικαστικό. Η κυρία Φαν Είναι πολύ σημαντικό. Καλό τους δύο συμπροέδρους να έρθετε σε επαφή με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων να βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Προέδρου έχει ικανοποιηθεί. Μπορούμε να κάνουμε την ακρόαση, να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, αλλά πριν αποτιμήσουμε τον υποψήφιο επίτροπο, θέλουμε γνωμοδότηση της νομικής επιτροπής για το ότι η αλλαγή του τελευταίες 72, συγγνώμη, ότι η δήλωσή του τις τελευταίες 72 ώρες έχει αλλάξει τρεις φορές. Αυτή είναι η αίτησή μου από πλευρά τη ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Πρόεδρος. Βεβαίω θα ελέγξουμε πριν την αποτίμηση. Και τώρα να σα εξηγήσουμε την ε, οργάνωση της ακρόασης. Ο υποψήφιος επίτροπος, ο υποψήφιος επίτροπος καλείται να κάνει μία εισαγωγική δήλωση. Στις προηγούμενες ε, ακροάσεις που έκανε η Επιτροπή Ήτρε είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε κι άλλε ακροάσει όπω ξέρετε, κάθε φορά η εισαγωγή ε, διαρκούσε 10 λεπτά. Για την Επιτροπή Περιβάλλον επίση ήταν 10 λεπτά. Αλλά θα σα δώσουμε λοιπόν 10 λεπτά. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, αν θέλετε να υπερβείτε τα 10 λεπτά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ισχύει και για τις άλλες ε, κοινέ ακρόασει. Κύριε Επίτροπε, θα έχετε 5 λεπτά επίση στο τέλος ε, τη ακρόαση. Κατόπιν, μετά την ε, παρουσίαση, θα υποβληθούν 45 ερωτήσεις. Ε, θα ακολουθήσουμε ε, τη διαδικασία ping-pong. Ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά απάντηση. Χωρίς συμπληρωματικές ερωτήσεις, επερωτήσεις. Δεν θα χωρίσουμε τις ερωτήσεις ανατομής πολιτικής ή κατά πολιτική ομάδα. ο χρόνος ε, ομιλίας ε, θα κατανεμηθεί με τους ίδιους κανόνες με τους, οποίες, με τους οποίους ε, λειτουργούμε στην Ολομέλεια. Σας παρακαλώ να τηρήσετε όλοι το χρόνο ομιλίας σας. Μόνο 5 δευτερόλεπτα ανοχή θα υπάρχει. Και 10 δευτερόλεπτα για σας κύριε Επιτρόπε. Μετά από αυτήν την μικρή υπέρβαση θα κόβω το μικρόφωνο θα βλέπετε το χρόνο σας και τους αστερίσκους όταν τον υπερβείτε στην οθόνη μπροστά σα Υπενθυμίζω ότι έχουμε ταυτόχρονη διερμηνία σε 23 γλώσσες. Μπορείτε λοιπόν να μιλήσετε και να ακούσετε τη γλώσσα σας. Σα σας παρακαλώ να μην μιλάτε υπερβολικά γρήγορα. Η συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης όλα αυτά εγγράφονται, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και εκ των υστέρων. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο